προστασία των θυμάτων της ε, τρομοκρατίας. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπιενκόφσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι έδειξαν για μία ακόμη φορά ε, την ριζοσπαστική σκληρή πλευρά της τρομοκρατίας. Γνωρίζουμε ότι πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια πολλές χώρες ήταν ο στόχος, η Ισπανία, η Εθνία, η Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Δανία. Η οδηγία του 2012 που άρχισε να ισχύει στα κράτη-μέλη τον περασμένο μήνα είναι το βασικό όργανο για τα δικαιώματα των θυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεσπίζει δεσμευτικούς κανόνες για όλα ε, τα θύματα της δημοκρατίας για προστασία και βοήθεια λαμβάνοντας υπόψη ε, τα μεμονωμένα δικαιώματα του κάθε θύματος αλλά δεν προβλέπει τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες αυτών των θυμάτων της τρομοκρατίας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αφορούν άτομα τα οποία πλήγησαν από αυτές τις επιθέσεις και έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Αυτά τα θύματα χρειάζονται ειδική προστασία ε, και βοήθεια που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους φυσικά που θα έχει σχέση με τη φύση αυτού του εγκλήματος. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισε η Επιτροπή ε, να θεσπίσει ειδικά μέτρα διατάξεις για αυτά τα θύματα ε, για την καταπολέμηση ε, της τρομοκρατίας. Αυτό στις 2 Δεκεμβρίου. Ο βασικός στόχος είναι να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις και όλα, όλα τα σχετικά σχετικές επιθέσεις όπως όμως και άλλες πράξεις όπως τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτή η πρόταση ανταποκρίνεται στην ανάγκη των θυμάτων της τρομοκρατίας, κυρίως η οδηγία αυτή ζητεί στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα θύματα ε, θα βοηθηθούν ε, με ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης προκειμένου να τους δοθεί και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να δίνεται όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Η Επίσης πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τα θύματα τρομοκρατίας η προτινόμενη οδηγία απαιτεί ότι αυτέ οι υπηρεσίε υποστήριξη να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι αξιόπιστε πληροφορίε. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ του, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλα τα θύματα τη τρομοκρατία είναι ενημερωμένα και λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι κανόνες για την υποστήριξη, τη βοήθεια ε, των θυμάτων δημοκρατίας ε, θα επουλώσει ε, τα τραύματα της οικογένειας και των θυμάτων και συνεπώς θα βοηθήσει όλη την κοινωνία. Επίσης υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωσης σχετικά σε όλα τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των, της ριζοστυπακοποίησης. Επίσης, στις 3 Οκτωβρίου φέτος άρχισε να λειτουργεί και χρηματοδοτήθηκε με 23 εκατομμύρια για την επόμενη τετραετία, ούτω ώστε ε, τα, άτομα, ε, τα αρμόδια άτομα επιτόπου να μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα. Ε, προέρχονται από πολλού τομεί αυτά τα άτομα, από την αστυνομία, από τι τοπικέ αρχέ, από τι φυλακέ, από κοινωνικού λειτουργού, από οργανώσει κοινωνία πολιτών, από δασκάλου και φυσικά πολύ σημαντικό από τι ομάδε και τι ενώσει των θυμάτων τη τρομοκρατία. Τα θύματα της Αξίζουν την αλληλεγγύη και τη βοήθειά μας. Επίσης, μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της ριζαστικοποίησης. Οι μαρτυρίες τους μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη. Επίσης, μία ομάδα εργασίας ε, για τη μνήμη των θυμάτων τρομοκρατίας συγκροτήθηκε. Θα βοηθήσει πολύ στην οργάνωση ε, της ημέρας ε, της ανάμνησης της 11 ε, η Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή κάνει μνημόσυνο για αυτά τα θύματα της τρομοκρατίας στις 11 Σεπτεμβρίου και θα την βοηθήσουν οι αρμόδιοι. Επίσης, αυτό γίνεται σε μνήμη όσους επλήγησαν και όσους εξακολουθούν να πλήττονται. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι οι φωνές των θυμάτων ακούγονται παντού, κυρίως μεταξύ των νέων, διότι ο πόνος αυτών των ατόμων δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθεί. Αυτά τα άτομα που είναι έτοιμα ε, να ακολουθήσουν τον εξτρεμισμό, έτσι θα σκεφτούν δύο φορές. Είμαι πεπισμένη ότι ο ρόλος αυτών των θυμάτων είναι πολύ σημαντικός. Θα φροντίσουμε ώστε οι ιστορίες τους και η εμπειρία τους να έχουν θετική επιρροή στα άτομα που κινδυνεύουν ε, να ε, μπουν σε ομάδες ριζαστικοποίησης. Ευχαριστώ. Uh, Περνάμε στου εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η κυρία Χιμένεθ Μπεσερίλ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταστηθεί μα θα πρέπει αυτό όμως να το αποδεχθούμε άπαξ και έχουμε τη, τη, τους Βάσκους της ΕΡΤΑ που σκότωσαν τον αδερφό μου και τη γυναίκα του. Οπότε δεν έχει σημασία από πώς έγινε. Δεν έγινε ότι ε, τώρα κάποιος πυροβολάει επειδή θέλει ανεξάρτητη χώρα των Βάσκων ή θέλει Ισλαμικό κράτος. Αλλά είδατε ε, τι έγινε στη χώρα μου και πόσο αξίζει γεγονός ε, αθώο. Έχουμε λοιπόν στο Ισπανικό κράτο το οποίο προθεί να καταπολεμήσει τον, ε, την τρομοκρατία και επομένω θα πρέπει αυτό ο αγώνα να είναι σύμβολο τη δημοκρατία κατά τη τρομοκρατία των τρομοκρατών. Έχουμε το σχετικό νόμο που δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα υλικά αλλά και σε θέματα ηθικά. Έχουμε επομένω την τρομοκρατία που χτυπήσει όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά αυτού του είδου ε, τις προβλέψεις που επιτέλους κάνουν κάτι για το θύμα και μόνος χρειάζεται τώρα να υπάρξει ε, αυτού του είδους το ε, νομοθετικό πλέγμα και πριν πρώτα πρώτα δικαίωμα στην προσοχή στη δικαιοσύνη, στην Αθήνα, στην αλήθεια, στην μνήμη επίσης. Η κανείς δεν θέλει να ωφελείται από όλα αυτά ένας τρομοκρατάτης και επίσης όλα αυτά σας τα λέω γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο συνεχώς προτείνει το να υπάρξει ένα ψήφισμα που να εγκριθεί για τα θύματα της τρομοκρατίας. Και έχουμε προσπαθήσει, έχουμε προτείνει κάτι για το πέριψη διάσκεψη των Προέδρων. Η ECR το ήθελε αυτό, αυτή την απόρριψη, όμως τώρα κάναμε ένα πρώτο βήμα. Οπότε βέβαια ε, αξίζουν τα θύματα μια οδηγία που να εγκριθεί από τα τρία θεσμικά όργανα και επομένως από τα δάκρυα να περάσουμε στις πράξεις και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν ε, από την τρομοκρατία, από τα θύματα. Κυρία Επίτροπε, πότε θα έχουμε την σχετική οδηγία. Δώστε μας μια ημερομηνία. Δέχεστε μια περώτηση από τον κύριο Σάλη. Επαναλαμβάνω. Από τον κύριο Σάνι. Δέχεστε περώτηση ή όχι. Ναι ή ου, ξαναρωτάει ο πρόεδρος. Η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ. Ναι, λέει. κυρια χιμενα μπεθεριλ ναι λεει εχετε τον λόγο, κύριε Σάνι. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφε, βεβαίως και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ε, για τον χαμό των μελών της οικογένειας σας όπως μας ε, αναφέρατε. Ξέρετε, στην πατρίδα μου την ε, Ουγγαρία ήμουν βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην περιοχή μας είχαμε πάρα πολλά θύματα των Ναζί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλούς νεκρούς. Παρακαλώ να πείτε στο κόμμα σας τι κάνουμε. Τι κάνουμε, κάνουμε διάφορα μέτρα τα οποία θέλουμε να πάρουμε από το κόμμα Φίντες για τα θύματα του Δευτέρου Πολέμου. Θέλετε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, τώρα συζητούμε για τα θύματα της τρομοκρατίας. Δεν μιλούμε για τους νεκρούς του πολέμου. Για μένα θα πρέπει όλα τα θύματα βέβαια να τύχουν τις ίδιες υποστήριξης, χωρίς καμία εξαίρεση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση. Δέχεστε τον κύριο Μπόγκοβιτ. Όχι. Μάλιστα. Ναι ή όχι it's misunderstanding i um, uh, Από τους Κυρία Κινίτση. Ενάμιση λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι τελευταίες τρομαδικές ε, επιθέσεις ε, μας ξαναθύμισαν ε, ότι κατεπήγεται ότι θα πρέπει τώρα να προσέξουμε ότι να μην κάνουμε κάτι μόνο για τους ε, δράστες, αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε προληπτικά. Αλλά και θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τα θύματα άμεσα ή έμεσα. Έχουμε το πρόγραμμα του 2009 της Στοκόλμης. Αναγνώριζε το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η σχετική νομοθεσία και τα μέτρα υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων αυτών των εγκλημάτων. Και βέβαια προτεραιότητα στα θύματα της τρομοκρατίας. Σε αυτή την κατηγορία καλύπτονται και οι συγγενείς των αμέσων θυμάτων. Και έχουμε την οδηγία του 29 του 2012 για τα θύματα εγκλημάτων και ανεγνώριζε εκεί ότι τα θύματα της τρομοκρατίας ε, είναι θύματα κάποιων εγκλημάτων κατά όλες τις κοινωνίες και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Σήμερα περισσότερα από πάντοτε θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει κάποια αλληλεγγύη, ε, θα, πώς θα υπάρξει κάλυψη εθνική και διεθνής ακριβώς όπω μας τα είπε σήμερα η κυρία Επίτροπος και την ευχαριστώ για την εισήγησή τη όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε υποστήριξη κοινωνική, υλική, ψυχολογική, ιατρική, ε, μακρόπνοη υποστήριξη για όσα υπέστησε. Γιατί υπάρχουν ε, ζημίες και υλικέ και ψυχολογικές ε, για τα θύματα της οικογένειας τους. Οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε το πώς θα υπάρξει νομική βοήθεια, να μπορεί κάποιος να ξαναστηθεί στα πόδια του και να υπάρχει επίση για τι ζημίες κάποια αποζημίωση και επίσης να αναγνωριστεί ο ρόλος των φορέων που βοηθούν και προστατεύουν τα θύματα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε εμείς κυρία Κίνητση, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, η σειρά. Τιμώθη Κέρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, η θλίψη μας ε, για αυτούς οποίους χάσαμε από την τρομοκρατία τα τελευταία έτη έχει πλέον καταγραφεί στην συνείδησή μας ε, ως ε, έθνη και ως ε, ένωση. Πρέπει πλέον να ξαναδούμε ποιον εμπιστευόμαστε και τι πιστεύουμε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η ρητορική του μίσους να δημιουργήσει νέα θύματα. Μετά τις αρχικές ημέρες του σοκ και της θλίψης είδαμε πώς επικράτησε η λογική και η συνοχή και βεβαίω η βαρβαρότητα του Ισλαμικού κράτους δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσει σε πράξεις ξένος. Θα νικήσουμε τον εχθρό και έτσι οι ζωές μας θα είναι χωρίς φόβο. Αλλά όχι με το τίμημα της ανοχής των θρησκειών που έχουν συνεισφέρει στην σημερινή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, του Άλντε. Η κυρία Παγκαζάρου Ορτουντουαρουής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι συνήθεις εγκληματίες συνήθως. Δεν θέλουν να διαφημίσουν τα εγκλήματά τους. Ούτε θέλουν να θεωρούνται ήρωες γιατί σκοτώνουν. Θέλουν να αποφύγουν, να γλιτώσουν τη δικαιοσύνη, άρα να μην είναι γνωστοί. Όμως, άλλος ονομαστή είναι τρομοκρατία. Όταν έχουμε σε δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή εγκλήματα τρομοκρατίας όπως η δική μας κοινωνία, που ε, χτυπάνε μικρούς και μεγάλους, γέρους, νέους, τους ε, κάνουν ανάπηρους, τους ε, βασανίζουν και θέλουν να χτυπήσουν, να διαλύσουν οι οικογένειες για να κάνουν μια προπαγάνδα. Και αυτό το οποίο θέλουν είναι να τρομοκρατήσουν όλο τον κόσμο, να πετύχουν κάποιες ε, αθέμητους σκοπούς. Θέλουν ε, να χτυπήσουν τις, τις χώρες, ακριβώς πως γίνεται και με τους τζιχαντιστές, θέλουν να αποδυναμώσουν τη δημοκρατία. Πρόκειται για κάποια εγκλήματα δημοσίου χαρακτήρα, είναι θύματα και ήρωες οι ε, δολοφόνοι αυτοί ε, και λένε ότι έχουν κάποια ικανότητα του να ελέγξουν την κοινωνία. Οπότε για αυτό το λόγο έχουν ε, διπλή φύση, ανθρώπινη και ιδιωτική. Τα θύματα θέλουν την ιδιωτική την βοήθεια γιατί τους έχουν σκοτώσει τους συγγενείς τους αλλά υπάρχει η πτυχή δημόσια γιατί και οι δημοκρατικές και κοινωνίες είναι οι στόχοι των τρομοκρατιών και γι' αυτό η δικαιοσύνη αλλά και η μνήμη χρειάζεται ε, χρειάζεται και είναι κάτι το απαραίτητο. Κανείς δεν θα τολμήσει να οδηγηθεί και ε, να πει ότι εγκρίνονται κάποια εγκλήματα όπως το που κάνουν οι τρομοκράτες κατά ανηλίκων και γυναικών. Αυτό όμως το κάνουν και κάποιοι ε, ζητούν ε, με συνενοχή και από φόβο να είναι ατιμόρυτοι οι τρομοκράτες. Και βέβαια τότε οι τρομοκράτες αισθάνονται περήφανοι το οποίο αυτό είναι αφόρητο. Τα θύματα υποφέρουν, χάνουν την αξιοπρέπειά τους και με κάθε τρομοκρατική προσπάθεια έχουμε περισσότερα θύματα και συνεχίζεται επομένω το έργο αυτών των τρομοκρατών και αυτό δεν τελειώνει τον κύκλο του ε, αίματος. Θεωρώ ότι εμείς υποφέρουμε στην Ισπανία με τρομοκρατία και το Κοινοβούλιο δεν έκανε ό,τι θα μπορούσε. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια συγκεκριμένη ε, οδηγία η οποία θα ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την ε, η κυρία Άντερσον για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ. Μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών και ετών θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την συμπαράστασή μου στα θύματα και τις οικογένειες του Το Ισλαμικό κράτος είναι ένα τέρας ε, του Φραγκενστάιν και τα κράτη-μέλη πρέπει να το σταματήσουν και για να το σταματήσουμε πρέπει να μην δέχονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, τα έσοδα που υπολογίζονται σε 2 εκατομμύρια την ημέρα από το ε, λαθρεμπόριο του πετρελαίου και βεβαίως να καλύψουμε και τις ανάγκες των εκατομμυρίων προσφύγων λόγω του τρόμου που ζουν ο βίος εξτρεμισμός έχει αυξηθεί σε μέρη τα οποία έχει τσακίσει, έχουν τσακίσει οι δυτικοί στρατοί και έτσι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος και βλέπουμε πως κλιμακώνεται η κατάσταση στην Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νέο μοντέλο επίλυσης διαφορών. Το να ρίχνουμε βόμβες δεν είναι η λύση. Στην Ιρλανδία το Βρετανικό κράτος σκότωνε ατιμόρυτα το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κύριος Νίκος Μιουσνιέκ, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λέει πως υπάρχει ουσιαστικά ατιμορρησία για το Βρετανικό κράτος. Δυστυχώς σε αυτές τις συζητήσεις δεν περιλαμβάνεται η κρατική τρομοκρατία. Και αυτά τα οποία ακούμε από το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία Σημαίνει πως θα πρέπει να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να καταδικάσουμε όλες τις πράξεις τρομοκρατίας ως ε, κράτος μέλος ε, και συμβαλόμενο μέρος ε, της ΕΣΔΑ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρεί το άρθρο 2 για το δικαίωμα στη ζωή σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τους πράσινους ο Ιαν Φίλιπ Άλμπρεχτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ πως όλοι σοκαριστήκαμε από τα θύματα της τελευταίας τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι και θεωρώ πως όλοι συμφωνούμε πως ε, το σοκ αυτό και ο τρόμος από τις επιθέσεις αυτές ε, πρέπει να μας ενώσει για να προστατευτούμε από τις επιθέσεις ε, και από το γεγονός πως η προστασία των θυμάτων δεν σημαίνει ότι πρέπει απλά να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικέ τους ε, ανάγκες αλλά και να προστατευτούμε από νέες ε, επιθέσεις για να μην έχουμε νέα θύματα. Θεωρώ όμως πως θα πρέπει να συγκεντρώσουμε και τα γεγονότα, τα στοιχεία που έχουμε στην ε, διάθεσή μας ε, για να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον και να μην κάνουμε στις πλάτες τους μια συναισθηματική συζήτηση και συναισθηματική αντίδραση. Αυτό ισχύει και όταν μιλάμε για τις αιτίες ε, της τρομοκρατίας που αν τις δούμε προσεκτικά στην ε, κρίση, βρίσκονται στην κρίση στη Μέση Ανατολή και στους εκεί πολέμους ε, που πρέπει να λύσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο γεγονός πως ε, πολλοί από αυτούς τους δρομοκράτες ριζοσπαστικοποιήθηκαν στην Ευρώπη και στις φυλακές της Ευρώπης. Πρέπει να τελειώσει αυτό και η ριζοσπαστικοποίηση αυτή να σταματήσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα γεγονότα, πώς θα είμαστε πιο ασφαλείς. Είναι σαφές, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών, καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και να μην έχουμε μια γενική παρακολούθηση όλων των πολιτών συλλήβδεν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το πρώτο καθήκον οποιοδήποτε κυβέρνηση είναι να αποδέχεται αυτό που θέλουν οι πολίτε. Λέγεται συχνά δεν μπορεί ποτέ να νικήσει η τρομοκρατία, αλλά αυτό δεν είναι αληθέ. Μπορεί να νικήσει όταν ένα μεγάλο αριθμό του κοινού ε, με συμπάθεια βλέπει το μακροχρόνιο στόχο τους. Αυτό χάρη το ζήσαμε τη Βόρεια Ιρλανδία. Λίγοι ε, παραδέχονταν ότι υποστηρίζουν τον IRA και τη το πολιτικό του σκέλος. Η τρομοκρατική απειλή έρχεται από τους φονταμεταλιστές, τους Ισλαμιστές που θέλουν ένα χαλιφάτο του Ισλάμ υπό την Σαρία. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι μας λένε είναι φιλερινικοί και μη βίαιοι, το δέχομαι. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα η, η πλειοψηφία, η μειοψηφία είναι το πρόβλημα και έχουν την ίδια θρησκεία. Τα διδάγματα της θρησκείας είναι ασυμίβαστα με τη δημοκρατία του δυτικού πολιτισμού. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την φονταμενταλιστική ιδεολογία στην κοινωνία μας. Είχα πει το περισμένο μήνα το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσουμε μια για πάντα όλη τη μαζική ε, αποχώρηση, μετανάστευση από Ισλαμικές χώρες. Το να υπάρχουν εκατομμύρια μετανάστες από Ισλαμικές χώρες ε, σημαίνει ότι παίζουμε ρωσική ρουλέτα με τη ζωή των πολιτών μας. Thank you. Um, so πολύ. Okay. Uh, blue card, I understand. Point of order, please. The point of order on the, on the rule. Διαδικασίες για τον κανόνα 11.2. Δηλαδή, τα μέλη πρέπει να χαρακτηρίζονται με ε, αμοιβαίο σεβασμό ως μέλος του Συνφέιν και επειδή έχω εκλεγεί στη Βόρεια Ιρλανδία από 160.000 άτομα που με ψήφισαν θεωρώ ότι δεν επιτρέπεται κάποιος αυτή την ε, αίθουσα να κάνει αυτή τη διασύνδεση που έκανε. Η ο τους του Σιν αγωνίστηκαν για μα με βάση την εντολή τους για να πούμε πώς θα εκπροσωπήσουμε το λαό μας και με βάση αυτό το πρόγραμμα το οποίο του παρουσιάσαμε. Περίπου μισό εκατομμύριο άτομα ε, στην Ιρλανδία αγωνίστηκαν για το Sinn Féin. Με βάση λοιπόν τον κανόνα 11.2 ε, το μέλος θα πρέπει να συμπεριφέρεται ε, με αμοιβαίο σεβασμό και δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο από ένα μέλος αυτού του Κοινοβουλίου. Thank you. Um, Μη εγγεγραμμένος ο κύριος Φουντούλης σήμερα η επιτροπή μας λέει πως ζητά προστασία και υποστήριξη για τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. πρέπει να απαλύνουμε τον πόνο των θυμάτων και των οικογενειών τους να αποφευθεί η ηρωοποίηση των τρομοκρατών να αναδειχθεί η αλήθεια και να θεσπιστούν ημέρες μνήμης για τα θύματα. δυστυχώς κάποιες χώρες της ένωσης έχουν διαφορετικά κριτήρια σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις ανάλογα με την ταυτότητα των θυμάτων και των δραστών και κυρίω ανάλογα με τις ιδεολογικέ του το ελλαδικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει και να παράσχει οποιαδήποτε μορφή στήριξη σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων όταν είναι έλληνες εθνικιστές. στις δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν γίνει εναντίον του κινήματός μας στο λαϊκό σύνδεσμο χρυσή αυγή με αποκορύφωμα την άνανδρη ψυχρό δύο μελών μας του γιου μου γιώργου φουντούλη και του μανώλη καπελώνη και τον βαρύτατο τραυματισμό του αλέξανδρου γέροντα το κράτος όχι μόνο δεν συμπαραστάθηκε στα θύματα και τις οικογένειές του ως όφιλε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία δύο χιλιάδες δώδεκα αλλά αντιθέτως συνεχώς προβάλλει εμπόδια αδιαφορεί και κολυσιεργεί. καταγγέλλω ότι σε πάνω από ογδόντα επιθέσεις δεν έχει γίνει ποτέ ούτε μία σύλληψη καλό λοιπόν θα ήταν αν η επιτροπή ενδιαφέρεται πραγματικά για τα θύματα να φροντίσει ώστε να προστατεύονται και να τιμούνται σε όλα τα κράτη ανεξάρτητα από την ιδεολογία τους. σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Τώρα, κυρία Βαζενμπεργκ, Βαζενμπεργκ χαίρομαι γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε ότι η οδηγία 29 του 2012 δεν μπορεί να καλύψει τα θύματα της τρομοκρατίας γιατί αφορά σε θύματα από εγκληματικές πράξεις. Η τρομοκρατία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι εξειδικευμένη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανθρωπότητα και τα θύματα και οι οικογένειές τους θέλουν ειδική ρύθμιση, θέλουν αναγνώριση και σεβασμό των δικαιωμάτων τους, κοινωνική, οικονομική, πολιτική, ψυχολογική, νομική στήριξη γιατί ανεξάρτητα αν οι δράστες είναι ψευτοεπαναστάτες που χτυπούν τους θεσμούς της δημοκρατίας όπως τη δικαιοσύνη το κοινοβούλιο την επιχειρηματικότητα το στράτευμα το πολίτευμα όπως έγινε στην πατρίδα μου με τη 17 Νοέμβρη που περιθωριοποίησε τη χώρα επί 30 χρόνια ανεξάρτητα αν είναι παρανοϊκοί που διακατέχονται από θρησκευτική ιδεοληψία όπως η Άισις δημιουργούν θύματα αίμα και πόνο και πανικό για τα δικαιώματα των οποίων χρειάζεται και απαιτεί η ειδική ρύθμιση. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η απάντηση της ευρωπαϊκής ένωσης στην τρομοκρατία πρέπει να είναι με περισσότερη δημοκρατία. η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η έλλειψη του φόβου και του πανικού διότι μόνο με τη θωράκιση των θυμάτων που είναι ήρωες σε αυτή την υπόθεση θα μπορέσει η τρομοκρατία να λάβει μια απάντηση με δημοκρατικούς κανόνες. σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, E Ο κύριος Χουάν Λόπες Αγγιλάρ. μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Ε, στις 13 Νοεμβρίου συνετάραξαν οι τρομοκές ενέργειε, αλλά πριν είχαμε και άλλε ενέργειε στο Σαλί και στο Λονδίνο το 2006, αλλά και στην Ισπανία η σφαγή του 2004 ε, μίλω ισπανικά, εκπροσωπώ την ισπανική κοινωνία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ξέρετε ότι εμά μας έχουν κατασφάξει, έχουμε ματώσει τόσα χρόνια από την ΕΤΑ και σας μιλώ εκ μέρους ενός κόμματος του Σοσιαλιστικού που έδωσε μακρά μάχη κατά της τρομοκρατίας και θέλουμε να θεωρείται κάτι υπερκομματικό κατά της τρομοκρατίας αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ζημία βάρος των θυμάτων για την αξιοπρέπειά τους, για την δικαίωμα στη δικαιοσύνη, για αποζημίωση των θυμάτων. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να βάλω το λιθαράκι μου για να βρεθεί τελικά μια ε, οδηγία ε, πέραν των όσων θεσπίστηκαν το 2012, τα οποία δεν καλύπτουν 100% την ιδιοτυπία ε, του πλήγματος κατά αυτών των θυμάτων. Γιατί υπάρχουν θέματα ε, πρακτικά, υπάρχουν θέματα ψυχολογικά, θέματα κοινωνικά, σε σχέση με τη δουλειά τους. Θα πρέπει επομένως να βρεθεί η σωστή θέση τους σε κάποιες διαδικασίες ε, ούτω ώστε να καλυφθούν αυτά τα χτήματα ε, της ε, τρομοκρατίας. Άρα χρειάζεται μια ειδική ad hoc οδηγία, ώστε να υπάρξει η ειδική αντιμετώπιση και αποζημίωση που χρειάζονται αυτά τα θύματα. Οπότε άπαξ και οι τρομοκράτες χτυπάνε κάποιους, να μην έχουμε μόνο τον πόνο και το αίμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το τι γίνεται με τον εκφοβισμό που προκαλούν οι τρομοκράτες. Άρα θα πρέπει παντού στην Ευρώπη να προστατεύσουμε τα θύματα. Παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, ένα Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να αναφερθώ στα πιο ευάλωτα θύματα, όπως παραδείγματος χάρη άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν τα άτομα αυτά στην πρώτη και σε επόμενες επαφές τους με αστυνομία και δικαιοσύνη να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη κάτι το οποίο σημαίνει συγκεκριμένα ότι ένα κοφό άτομο θα πρέπει να έχει έναν διερμηνέα κοφών στην ανάκριση και στο δικαστήριο. Ένα άτομο το οποίο έχει νοητική υστέρηση θα πρέπει να έχει ένα άτομο της εμπιστοσύνης του μαζί. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη. Αυτό εξακολουθεί να μην συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι το δικαίωμα του να καταλαβαίνει κανείς και να γίνεται αντιληπτός και θα πρέπει να εφαρμόζεται. Thank Σας ευχαριστώ. Νίκολσον για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εκφράζω τη συμπάθειά μου για όλους όσοι υπέφεραν από την τρομοκρατία στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης και κυρίως ε, στην Βόρεια Ή Ιστορικά οι τρομοκράτες μοιράστηκαν την εμπειρία τους και τη γνωσία τους μεταξύ των ομάδων Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς ε, να ανταλλάσσουμε εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Οι επιβιώσαν της τρομοκρατίας ε, χρειάζονται υποστήριξη πολύ μετά ε, το πλήγμα. Γι' αυτό τα άτομα, οι οικογένειες, οι κοινωνίες θα πρέπει να βοηθηθούν μετά από την τρομοκρατική επίθεση. Είναι περίπλοκα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και χρειάζονται πολύ χρόνο. Οι επιζήσαντες έχουν το δικαίωμα στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη και στο να μην έχουν τραυματιστεί από τους τρομοκράτες που δοξάζουν τις τρομοκρατικές τους πράξεις. Υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ των αθών θυμάτων ε, και των δραστών θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα θύματα και όχι τους δάστες. Uh, Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εδώ. Χαιρετίζω αυτή την πρόταση και θέλω να συγχαρώ ε, τον συνάδελφο για τη δουλειά που έχει γίνει υπογραμμίζοντα τι ανάγκε που έχουν τα θύματα σε όλε τι κοινωνίε. Όπω είπαν οι προραλήσαντε, έχουμε ευθύνη να βοηθήσουμε τα άτομα που είναι αθώα θύματα τη τρομοκρατία σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στη χώρα μου την Ιρλανδία, ε, αντιμετωπίσαμε μια παράνομη καμπάνια από το IRA και άλλες οργανώσεις που σκότωσαν, εκφόβησαν και κυρίως εξασφάλισαν ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα τους για άλλες δραστηριότητες. Έχουμε την ευθύνη να υποστηρίξουμε τα άτομα που έχουν να αντιμετωπίσουν απώλειες, θύματα, λύπη. Η χώρα μας πέρασε μεγάλες αλλαγές ε, μετά από τη συμφιλίωση. Ε, πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα τώρα, απευθύνομαι στην Επιτροπή. Και πρέπει να δούμε σε έξι μήνες κατά πόσον σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μεταφέρει την νομοθεσία και καλό την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί πολλά πρέπει να γίνουν. It's really late, but, uh, maybe Mr. Nicholson... Αλλά ίσως ο κύριος Νίκολσον θα δεχθεί να απαντήσει. Να απαντήσει η κυρία Χιμερές Περίελ. Yes. Ε, ε, ναι, ναι, ναι, λέει η κυρία Μπεφερίλ. Συμπαθάτε με, συμπαθάτε με, πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να ρωτήσω τίποτε τον κύριο Νίκολσον. Απλώς αυτό το οποίο θέλω είναι να μου δώσετε μισό λεπτάκι για την συζήτηση που αφορά τα θύματα, για να θυμηθούμε αυτούς που δύο μέρες πριν ε, πέθαναν και σκοτώθηκαν στην Καμπούλ, στην Ισπανική πρεσβεία. Είναι δύο αστυνομικοί που προστάτευαν αυτή την πρεσβεία ή στην Καμπούλ και αξίζει να τους θυμηθούμε ή αυτή τη συζήτηση για τα θύματα της τρομοκρατίας. Uh, I understand you, I can δεν ήταν ερώτηση βεβαίως αυτό. Έτσι, η μπλε κάρτα είναι μόνο για ερωτήσει. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τις αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις του Ντάις στο Παρίσι, με τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στην αποφασιστική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στην προστασία των θυμάτων της εκφράζουμε λοιπόν τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης του ντάεσ. η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας 29 του 2012 στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ανοίγει ένα πρώτο πεδίο προστασίας των θυμάτων της τρομοκρατίας. όμως δεν είναι αρκετό γι' αυτό απαιτείται η θέσπιση νέας οδηγίας ειδικής για την προστασία και την βοήθεια των θυμάτων της τρομοκρατίας ιδίως μετά τις μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις των τζιχαντιστών και αυτό είναι πλέον μια αναγκαιότητα η θέσπιση αυτής της οδηγίας. για να αντιμετωπιστούν όμως καλύτερα τα και να υπάρξει προστασία των θυμάτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά η τρομοκρατία. ειδικότερα όσον αφορά την τρομοκρατική δράση του ντάεσ θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της τουρκίας και όσων αραβικών χωρών στηρίζουν τον ντάεσ στην τουρκία Συρία. Επιπλέον πρέπει να εμπεδοθεί η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τρομοκρατική απειλή για όλο τον κόσμο και οι ιδιομορφίες των εγκλημάτων που ε, γίνονται και η σημασία όσων παθαίνουν τα θύματα μας κάνουν να μην ξεχνούμε το ότι χρειάζεται μια οδηγία σύγκεξης για αυτό το παγκόσμιο καινούργιο ε, φαινόμενο το οποίο τώρα έχει αλλάξει. Θα πρέπει επομένω να προσέξουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να καλύψουμε καλύτερα τους πολίτες. Να μην έχουμε ε, γραφειοκρατία όσον αφορά την πλαισίωση αυτών των θυμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια βιώσιμη και θα πρέπει η προστασία αυτή να είναι διασυνοριακή. Χρειάζονται συμπάθεια, ανθρωπιά, χρειάζονται κατανόηση, αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικέ οι σχετικέ αρμόδιε υπηρεσίε να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα και τους εγκληματίες. Αυτό να γίνει με τις υπηρεσίε πληροφοριών, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτούς που κατά τύχη έγιναν θύματα. πρόκειται για κάποιους που θέλουν ολοκληρωτισμό και θέλουν να καταστρέψουν την ελευθερία μας και τον τρόπο ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ. Προσφάτως χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα αντί να βλέπουμε τα θετικά θέματα που βελτιώνουν το μέλλον της νεολαίας μας. Χρειάστηκε να ασχοληθούμε με την τρομοκρατία, με τις συνέπειες της τρομοκρατίας και πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση των θυμάτων. Βεβαίω, ελπίζουμε ότι όλα τα μέτρα που διαθετήσουμε θα είναι αποτελεσματικά και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην πρόληψη αυτών των επιθέσεων. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι επιζήσαντες των τρομοκρατικών επιθέσεων έχουν λυγεί για όλη τους τη ζωή και οι οικογένειε του, Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πρώτον για να προλαμβάνουμε αυτέ τι επιθέσει, αλλά και αν συμβούν θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο προσπαθώντας ε, να παράσχουμε ως τον ετών μεγαλύτερη βοήθεια με όλους τους οργανισμούς που έχουν, να τους ε, παράσχουμε και ψυχολογική βοήθεια σε αυτούς και στην οικογένειά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη αναμφίβολα είναι η ήπειρος της ανοχής. Δυστυχώς αναμφίβολα επίσης η Ευρώπη είναι και ήπειρος που υπάρχει τρομοκρατία. Μπάτεν Μάχοφ στην Ιταλία, ΑΕΡΕΙ στην Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο και πρόσφατα στο Παρίσι, όλες έλαβαν χώρα στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο η οδηγία αυτή είναι απαραίτητη. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη με τα θύματα της τρομοκρατίας και πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτά τα θύματα της τρομοκρατίας επειδή αυτά τα άτομα ζουν κάπου, σε ένα χωριό, σε μια πόλη. Θα πρέπει να ε, συνδράμουν όλες οι υπηρεσίες γιατρικές, κοινωνικές και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω θερμά αυτή την οδηγία. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μου δώσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ο 20ος αιώνας ε, σημαδεύτηκε με διάφορα, από διάφορα πολιταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν αναγνώριζαν δικαιώματα στους ανθρώπους ε, αλλά και Ήδη στον 21ο αιώνα έχουμε ομάδε που επιτίθενται σε άμαχου, ε, αλλά είναι διαφορετικές από τις παλες Τώρα έχουμε μαζική τρομοκρατία, εννοώ μαζικές επιθέσεις. Και αυτές οι επιθέσεις ε, πραγματικά πηγαίνουν ενάντια στην ε, δημοκρατική μας κοινωνία και είναι πάρα πολλά και τα θύματα αυτών των επιθέσεων. Γι' αυτό στηρίζω την πρόταση που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή. Πρέπει τα θύματα να τα προστατεύσουμε αλλά και να προλάβουμε και τις αιτίε των τρομοκρατικών επιθέσεων. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Επιτροπός, κυρία Πινιακόφσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα διαβιβάσω οπωσδήποτε το πνεύμα της συζήτησης αυτής, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ τα θέματα της δημοκρατίας και της ρίζοσπαστικοποίησης και σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας για την πρόληψη της ρίζοσπαστικοποίησης που εγκρίνατε πριν από λίγες εβδομάδες και βεβαίως ε, αυτό θα πρέπει να γίνει ε, στο τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία των διαφόρων φορέων που βρίσκονται επί τόπου για να στηρίξουμε και τους, ε, τα θύματα της τρομοκρατίας και της οικογένειάς τους. Η Κομισιόν αναγνωρίζει την διαφορετική κατάσταση των θυμάτων της τρομοκρατίας σε σχέση με την υπόλοιπη εγκληματικότητα. Γι' αυτό προτείνουμε τη νέα αυτή οδηγία και βεβαίω έτσι θα στηρίξουμε και τα θύματα και τι οικογένειε του και περιμένουμε και την δική σα στήριξη του Κοινοβουλίου για να εγκριθεί γρήγορα η προτινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση τη θερμοκρατία. και βεβαίω θα διαβιβάσω το μήνυμα στην Επίτροπο Γύρωβα για το έτοιμά σα ε, για να δούμε πότε θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε κύριοι. Τελείωσε η συζήτηση. Και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουμε την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο